Okay. I think we are all set. Είμαστε έτοιμοι. Πρώτο σημείο, μία ψηφοφορία για την έγκριση ένστασης για το γενετικά, τον γενετικά τροποποιημένο αραβόσιτο. Ψηφίζουμε μία φορά ηλεκτρονικά, άρχεται ψηφοφορία. Did everyone vote? Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο σημείο, αντίρρηση για το τρίτον X100. Μία ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Περνάμε σε άλλη μία ψηφοφορία, δεύτερη ανάγνωση για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενη ψηφοφορία. Δεύτερη ανάγνωση και πάλι. Κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και την τροποποίηση τη Οδηγία 2001 κάθετο 83, του Κανονισμού 178 κάθετο 2002 και του Κανονισμού 1223 κάθετο 2009. Μία ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενη ψηφοφορία, σύμβαση της Μιναμάτα για τον Ιδράργυρο. Υπάρχει συνένεση, μία είναι η ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Επόμενο σημείο, εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα ορχείων. Ψηφίζουμε το σχέδιο έκθεσης του κύριου Χολβένη. Τροπολογία 14 λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας.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 Ναι, μάλιστα. Μπορεί να είμαστε κοντά στις θετικές και αρνητικές ψήφους. Πέρας. Μία. Για μία ψήφο. Νομίζω πως κάποιος δεν ψήφισε αυτή τη φορά σε σχέση με αυτούς που ψήφισαν την προηγούμενη τροπολογία. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40. Υπέρ. Κατά.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 Πέρας. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια στον κύριο Χολβένη. Επόμενο σημείο. Γνωμοδότηση για τα μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της Σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη διατήρηση των θηνοειδών του Ατλαντικού. Δεν υπάρχουν συμβιβαστικές τροπολογίες. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τροπολογία 7. Ποιος είναι υπέρ. Σας ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Την τροπολογία 9. Ναι. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε την 37. Εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τι σας είπα. Α, 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, Ξανά, 41. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 40. 2, 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται.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 Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. 17. Άρχεται η ψηφοφορία και πέρας. Εγκρίνεται. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ.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 απορρίπτεται. 1 υπέρ, κανά, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε την 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Δεν σηκώνατε τα χέρια. Ας ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία για την γνωμοδότηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια στην κυρία Μπριάνο. Επόμενη. The next item is... Επόμενο σημείο. έκθεση του κ. Πατριτσέλο για τη χορήγηση εγγύηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικέ δραστηριότητε που υποστηρίζουν επενδυτικά έργα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 25 και 34 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 30 υπέρ, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά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 εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία για τη γνωμοδότηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία. Και έχουμε πολύ χρόνο. Τελειώσαμε για το πρωινό. Οπότε θα τα ξαναπούμε στις 3 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.